στην έκθεση της κυρίας Γκαρντίνη τώρα. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Δίνω τον λόγο στη συνάδελφο κυρία Γκαρντίνη ως εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι σήμερα για όλους όσους έχουν εργαστεί γύρω από το θέμα αυτό έχει φτάσει μια σημαντική μέρα, συγκινητική μέρα. Υπήρξαν μακρότατες ίδια πραγματεύσεις και τελικά ο νέος μηχανισμός πολιτικής προστασίας σχηματίζεται. Είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα στην πορεία για μια Ευρώπη ασφαλέστερη, για ένα κόσμο περισσότερο ασφαλή. Να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου προς το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάστηκαν με επικοδομητικό τρόπο από την πρώτη στιγμή μαζί μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ακόμη φορά απέδειξε ότι είναι το ευρωπαϊκό όργανο που βρίσκονται πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες στην παρούσα φάση δεν ζουν την Ευρώπη με πολύ θετικό τρόπο και είναι κάτι που αφορά ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών μας. Υπάρχουν όμως κάποιοι χώροι ευρύτατοι στους οποίους η Ευρώπη εργάζεται και μπορεί να αποδείξει στους πολίτες ότι η Ευρώπη βρίσκεται κοντά τους, ότι η Ευρώπη είναι φίλη τους και ότι η Ευρώπη είναι ο κοινός χώρος των πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς εγγράφουμε ένα επιπλέον κεφάλαιο μέσω της αλληλεγγύης την οποία εκφράζουμε με τον νέο μηχανισμό που αλλάζει εντελώς την φιλοσοφία της πολιτικής προστασίας που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το χρήσιμο. Εμείς σήμερα λέμε στους συμπολίτε μας ότι η Ευρώπη είναι μαζί τους, είναι δίπλα τους. Έχουμε να κάνουμε με έναν δρόμο διαλόγου, με μια πορεία επικοινωνίας. Εγώ ξεκίνησα με μια θέση που στήριξε το Κοινοβούλιο εξ αρχής και μπόρεσα να εργαστώ κατά από συνθήκες καλές. Οι θέσεις μου αυτές ενισχύθηκαν για προς την κατεύθυνση της προστασίας ε, των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Και η Κρυσταλίνα Γεωργίευα έδειξε όλη της την ικανότητα και το πάθος της ε, βρίσκεται επιτόπου στα προβλήματα και ξέρει με ποιο πραγματιστικό τρόπο μπορεί κανείς να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές φροντίζει τους πολίτες, τις οικογένειές τους, τις ανθρώπινες αυτές καταστροφές και τα ανθρώπινα αυτά ερήπια που ε, είναι προϊόν της βίας της φύσης. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν με τις προτάσεις της να μην μεταφέρει αυτήν την πραγματική ανθρωπιστική αντίληψη για το θέμα που μας αφορά. Γράψαμε νέα κεφάλαια λοιπόν και για την πρόληψη και την προπαρασκευή. Πρόληψη. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες εξ αρχής. Θέλουμε οι καταστροφές να προλαμβάνονται. Εάν δεν προλαμβάνονται θέλουμε με ουσιαστικό τρόπο να μειώνονται οι επιπτώσεις τους, τα προβλήματα που δημιουργούν. Θέλουμε να προωθήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης σαν παράδειγμα προγράμματα διαχείρισης κινδύνων, βασικά προγράμματα για την σωστή ε, διαχείριση των προβλημάτων. Η δημιουργία του εθελοντικού πουλ μέσων, τη ομαδοποίηση των διαθεσίμων μέσων που θα επιτρέψει να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός σωστά. Εγώ δεν θα σταθώ στα τεχνικά, θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι έχουμε προσπαθήσει να ξεπεράσουμε τις, ε, τους δισταγμούς των κρατών μελών, προωθώντας και την αλληλεγγύη αλλά και την επικουρικότητα που διατρέχουν το σύνολο του κειμένου μας. Ε, σας ευχαριστώ και θα ακούσω τώρα και τις παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων. Ευχαριστούμε και κυρία συνάδελφε Γκαρντίνη. Για την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Επίτροπος Γεωργίευα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκουαρντίνη και όλους τους ευρωβουλευτές που συνεργάστηκαν ακούραστα επί χρόνια για να παρουσιάσουμε σήμερα από κοινού το νομοθεσία που συζητάμε. Το θέμα είναι καλύτερη προστασία για τους πολίτες μας και για τις οικονομίες μας. Γιατί υπάρχει μια τάση αύξησης των θεομηνιών και θέλουμε να υπάρξει και καλύτερη περίθαλψη υποβοήθηση των θυμάτων των θεομηνιών. Θα ξέρετε ότι τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίσαμε πολύ μεγάλη αύξηση της συχνότητας και της έντασης τέτοιων καταστροφών εδώ στην Ευρώπη. Ε, σε 10 χρόνια Χάσαμε 100.000 πολίτες λόγω καυσώνων, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών και επίσης επηρεάστηκε αρνητικά η οικονομία μας λόγω του κόστους άνω των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρατηρείται διεθνώς. Τα τελευταία τρία χρόνια και μόνο και για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το κόστος, οι ζημίες ξεπέρασαν 100 δισεκατομμύρια δαλάρια το χρόνο και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι όλο το κόστος γιατί δεν καλύπτει όλες τις ζημίες. Το περασμένο καλοκαίρι οι πλημμύρες έπληξαν ιδιαίτερα την κεντρική Ευρώπη και μας κόστισαν πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τη Γερμανία ήταν το υψηλότερο κόστος, η υψηλότερη ζημία που σημειώθηκε ποτέ. Υπάρχει λοιπόν πραγματικά αυτή η τάση και με τη νέα αυτή νομοθεσία θέλουμε να κάνουμε ένα άλμα να δημιουργήσουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης των θεομηνιών με πρόληψη και προετοιμασία αλλά και προγραμματισμένα προγράμματα περίθαλψης. Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία τα κράτη-μέλη δέχονται τη νομική δέσμευση να προετοιμάσουν προγράμματα αντιμετώπισης και εθελοντικά να συνδυάσουν πόρους για άμεση αντιμετώπιση αν πλήξει κάποια χώρα μας κάποια τέτοια θεομηνία. Αυτή η νομοθεσία λοιπόν ανταποκρίνεται σε μια έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την έχω ακούσει και εγώ ίδια πολλές φορές ότι χρειάζεται, ότι πρέπει η Ευρώπη να αντιδράει ενωμένη σε τέτοιες θεομηνίες και το εργαλείο αυτό το ζητήσατε εσείς πολλές φορές. Τώρα θα γίνει πραγματικότητα. Ακολουθήσαμε μία προσέγγιση bottom-up. Δηλαδή βασιζόμαστε σε θελοντική συνεργασία των χωρών μελών με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Και τελειώνω δηλώνοντας ότι πριν από μερικές εβδομάδες στις Φιλιππίνες είδα με τα μάτια μου τι σημαίνει η ενωμένη δράση της Ευρώπης και είμαι πολύ περήφανη για αυτό που καταφέραμε εκεί. Στο μέλλον η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας θα απαιτεί και τη δική σας υποστήριξη στην οποία υπολογίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε Γεωργίευα. Ακολουθούν τώρα οι συγητές. Πάσκου, δεν παρίσταται. Συνάδελφε Στρίφλερ, έχετε τον λόγο. <clears throat> Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση απόφασης για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενισχύει σαφώς το πρόγραμμα συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις φυσικές καταστροφές και να βελτιώνει τις δυνατότητες παρέμβασης. Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία του συστήματος αυτού ε, εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες ε, του τρίτου κόσμου. 70% λοιπόν του προϋπολογισμού θα καλύψει τις ανάγκες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εδώ και πέρα και 30% μόνο στο εξωτερικό. Συνεπώς η συμφωνία για το δημοσιονομικό δεν, δεν είναι συμβατή, δεν συνάδει με την πραγματικότητα και με τις προσπάθειες βοήθειας στις χώρες που βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης. Ευχαριστούμε συνάδελφε Στρίφλερ. Ο κύριος Σταυρακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο μηχανισμό πολιτική προστασία έχει ανδιαφυσβήτητη προστιθέμενη αξία και αποτελεί μια ορατή, έμπρακτη και σημαντική έκφραση αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ του πολίτε τη, όπω για παράδειγμα με την ενεργοποίηση του μετά τον καταστροφικό σεισμό στην αγκύρα τη Ιταλία το 2009, αλλά και η ενεργοποίηση του μηχανισμού για τρίτε χώρε προσφέρει σημαντική ανακούφιση για την αντιμετώπιση καταστροφών σαν και αυτέ που προκάλεσε ο πρόσφατο τυφώνα χάιαν στι φιλιππίνε. όπω γνωρίζουμε η πρόληψη των καταστροφών είναι υψή τη σημασία και κοστίζει στον ευρωπαίο πολίτη πολύ λιγότερο από την αντιμετώπιση του. όσον αφορά τη χρηματοδότηση του μηχανισμού δεν μπορώ να μην εκφράσω την απογοήτευσή μου κύριε πρόεδρε για το τελικό ποσό που ανέρχεται στα 368,42 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις τόσο εντό όσο και εκτό τη ένωση για την επόμενη πενταετία μειωμένο από την αρχική πρόταση ύψου 513 εκατομμυρίων ευρώ. ωστόσο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αναγνωρίζει τι προσπάθειε εξορθολογισμού που καταβάλουν τα περισσότερα κράτη μέλη. για τον λόγο αυτό και για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπο τη υπάρχουσα ενίσχυση η Στούμε πολύ συνάδελφε Σταυρακάκη. Ξεκινήσαμε πολύ έγκαιρα στην ώρα μας και κάποιοι εισηγητές ακόμα και αν δεν παρίστανται. Τώρα ήρθε ο κύριος Πάσκου. Κύριε Πάσκου έχετε τον λόγο παρακαλώ. Πάσκου, Κύριε Πάσκου θέλετε να παρέμβετε. Ο μηχανισμός αυτός πολιτικής προστασίας είναι κάτι βασικό για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστροφών. Η Επιτροπή Εξωτερικών υποστήριξε τη γενική αυτή προσέγγιση που συνίσταται στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης αντί των μεμονωμένων ad hoc μέχρι τώρα μηχανισμών. Η Επιτροπή Εξωτερικών δέχεται αυτές τις ιδέες και τονίζει τη σημασία της ε, αξιολόγησης των κινδύνων εκ των προτέρων και την ανάγκη να υπάρχει συνεπής και ενιαία αντιμετώπιση και αυτό το βλέπουμε σαφώς στο έγγραφο που συζητούμε σήμερα. Στη γνωμοδότησή μας τονίσαμε ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης από τη μία και συνέπειας των ε, πολιτικής, ε, της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης από την άλλη. Υποστηρίζουμε λοιπόν την Επίτροπο Γεωργίευα στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε συνάδελφε Πάσκου. Ο κ. Λασάκη δεν παρίσταται οι τοποθετήσει από πλευρά κοινοβουλευτικών επιτροπών ολοκληρώθηκαν. Ακολουθούν οι αγορητές εξωμάτων των ομάδων. Ξεκινά ο κύριο Ζέμπερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας βλέπει κανείς πολύ καλά πως πρόσθετη αξία απορρέει και αναγνωρίζουν αυτό οι πολίτες στην Ευρώπη με την παροχή βοήθειας. Εδώ η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευδιάκριτο πρόσωπο και από κοινού πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη προς αυτό. Για μας ήταν σημαντικό στην κοινοβουλευτική μας ομάδα η αρχική αρμοδιότητα και υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλιστεί. Πρωτογενώς αυτά τα κράτη-μέλη να είναι αρμόδια όταν στην επικράτειά τους ή ανθρωπογενώς κιόλας υπάρχουν καταστροφές ε, Ωστόσο πάντα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις ε, που έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και διαστάσεις και είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι. Έχουμε ήδη τέτοια βιώματα στην Ευρώπη ότι μπορέσαμε να βελτιώσουμε το συντονισμό μας στη συνεργασία μας. Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, να κάνουμε το επόμενο βήμα, συγκεκριμένα να διαθέσουμε κονδύλια πράγμα το οποίο κάναμε ήδη. Και έτσι με πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και τη διάθεσή τους και τον επιμερισμό 70-30 ως κλείδα ευρωπαϊκά να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Έχει νόημα αυτό. Και είναι σημαντικό και από τα βιώματα, από την πείρα μας να συναγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα σε σχέση με την πείρα μας. Και καταδείχθηκε ότι υπάρχει μεγάλη πρόσθετη αξία όταν γοργά μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη και όταν επιμέρους κράτη-μέλη μπορούν έτσι να βοηθήσουν και να δράσουν αποτελεσματικά. Το σύστημα των προτύπων και τρόπων που δημιουργήσαμε έχει και αυτό νόημα, διότι έτσι μπορούμε να πούμε εδώ έχει ένα κράτος ειδικότητα σε αυτό και έτσι ο συντονισμός πανευρωπαϊκά κεντρικά πρέπει να επιτυγχάνεται αυτός ο συντονισμός ε, για την αλληλεγγύη. Σημαντικό είναι να μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη αν θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο α, όσον αφορά τα επιμέρους πρότυπα. Και όλα αυτά εδώ σε σχέση με τα θέματα επικουρικότητας από πλευράς των μελών είναι νομίζω ένα αναγκαίο λογικό βήμα ως συνέπεια να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα. Έχουμε πρώτη εμπειρία ήδη στι Φιλιππίνες. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Εντίτε Στρέλα από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντα την εισηγήτρια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, επίση προεδρίε, η ε, Ιρλανδική και Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου που κατέβαλαν προσπάθειες ώστε αυτή η συμφωνία να καταστεί εφικτή. <clears throat> και ξεκινώντας από τον Ιανουάριο 2014 να μπορέσουμε να έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει. Η συχνότητα των καταστροφών αυτών αυξήθηκε με ζημιές ε, σε μέσο επίπεδο ετήσιο περίπου 0,25% <clears throat> του ΑΕΠ παγκόσμια. Τα τελευταία 20 χρόνια οι θεομηνίες που σημειώθηκαν στην Ευρώπη ε, είχαν σαν συνέπεια 90.000 θύματα έπληξαν και κατέστρεψαν περιουσίες 29 εκατομμυρίων ανθρώπων και είχαμε και οικονομική απώλεια 211 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι αριθμοί που πρέπει να τύχουν της προσοχής μας. Μια ναι, και αναφέρθηκε και η τελευταία δραματική περίπτωση που έλαβε χώρα στις Φιλιππίνες. Τώρα λοιπόν αυτή η αύξηση και, σοβαρό... και του αριθμού και της σοβαρότητας των καταστροφών παγκόσμια αυτά οφείλονται όλα στις κλιματικές αλλαγές και σε επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Πράγμα που απαιτεί πολιτικές πρόληψης ως προτεραιότητα από πλευράς μας. Η συνθήκη της Λισαβόνας συμπεριλαμβάνει μια ρήτρα αλληλεγγύης και θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να βοηθούν το ένα το άλλο αμοιβαία σε περίπτωση θεομηνιών ή ανθρωπογενών καταστροφών <clears throat> και εντός και εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο και εδώ ε, με σημαντικό τρόπο τρόπο ε, την πρόταση, την φιλόδοξη πρόταση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με την θέση που ελήφθη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος κιόλας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ε, ε είμαστε ε, εκτός των πλαισίων του ευκταίου όσον αφορά το, τα, τις δικές μας φιλοδοξίες. Και βλέπουμε εδώ σε σχέση και με την κοινή θέση που υιοθετείτε, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι περισσότερο είναι, αξίζει να προβλέψουμε καταστροφές και να είμαστε στην πρόληψη αποτελεσματική παρά να διορθώνουμε τα, τις καταστροφές στο τέλος τέλος, να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάτι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Thank you, President. Member. Ο μηχανισμός προστασίας, πολιτικής προστασίας έχει σαν στόχο την κατανομή των προσπαθειών ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Όταν ένα κράτος μέλος έχει να αντιμετωπίσει μια θεομηνία, πλημμύρα, πυρκαγιές κτλ. τότε κινητοποιείται το κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από το αίτημα σύνδρομής του κράτους μέλους και των διεθνών οργανώσεων. Μέχρι τώρα ευτυχώς η χώρα μου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάστηκε να προσφύγει σε ένα τέτοιο σύστημα αλλά έχει ερευνήσει την δυνατότητα χρήσης του συστήματος αυτού αν δημιουργηθεί ανάγκη στο μέλλον. Η περιοχή μου παρουσιάζει κινδύνους, ιδιαίτερα ε, σε σχέση με το φαινόμενο της ε, πλημμύρας ε, και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα μια μικρή πόλη στην εκλογική μου περιφέρεια πλημμύρισε. Γι' αυτό λοιπόν η δυνατότητα λειτουργίας του μηχανισμού αυτού εξαίρει θα έλεγα τη σημασία του σωστού συντονισμού. Ο συντονισμός θα αποτρέψει το χάος και την κατασπασάληση των πόρων και των χρημάτων. Η αυξημένη προπαρασκευή, όπως επίσης και το λεγόμενο pooling, η ομαδοποίηση των μέσων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των συνεπειών των θεομηνιών είναι κάτι το θετικό. Μέσω διαπραγματεύσεων αποφύγαμε εμείς να ξεπεράσουμε κάποιες υπερβολικές, κάποια υπερβολικά επίπεδα δάπανων με σωστή ενημέρωση και σωστό προγραμματισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποσυρθούν σαν παράδειγμα από κάποιες ομάδες παρέμβασης ε, εθελοντικές λεγόμενες εφόσον αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι χώρες αντίστοιχα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Γκαρντίνη, η για την πολύ καλή συνεργασία. Αυτή η απόφαση όσον αφορά την πολιτική προστασία εναντί καταστροφών καταδεικνύει ότι σαφείς βελτιώσεις μπόρεσαν να επιτευχθούν πρώτον όσον αφορά και τα κονδυλία αλλά επίσης όσον αφορά τα θέματα της προετοιμασίας και του συντονισμού σωστικών δράσεων αυτό το έργο πρέπει ως προπαρασκευή για την και προσαρμογή μας στις κλιματικές αλλαγές να θεωρήσουμε τις συναφείς δράσεις και από πλευράς ασφαλιστικών εταιριών καταδεικνύεται ότι οι ζήμιες αυξάνονται διαρκώς και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, πυρκαγιές ε, το ε, φθινόπωρο είχαμε θύελες που έπληξαν το βορρά της Ευρώπης ε, και κατέστρεψαν πάρα πολλές περιουσίες. Η καλή προετοιμασία σε σχέση με όλα αυτά μπορεί να οδηγήσει στο να μειωθούν τέτοιου είδους επιπτώσεις και καταστροφές αν δράσουμε προληπτικά. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι δεν τα κατάφερε η βιομηχανία και επιχειρήσεις ε, να δράσουν αποτελεσματικά. Έχουμε υπόψη τα διάφορα ατυχήματα, βιομηχανικά ατυχήματα, την διαρροή ε, δηλητηροδών ουσιών ε, που το ένα οδηγεί στο άλλο και τελικά έχουμε καταστροφές. Και πρόσφατα είχαμε και σε μια αλουμινοβιομηχανία ένα ατύχημα. Κόκκινη λάσπη κατέληξε σε ποτάμια και πλημμύρισε χωριά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούσαν αυτά να είχαν αποφευθεί αν είχαν συντηρηθεί σωστά φράγματα και αυτό δείχνει ότι ε, η αποφυγή μεγάλων ατυχημάτων δεν είναι μόνο ε, θέμα μεγάλων σωστικών υπηρεσιών και δράσεων αλλά σωστής δράσης στο επίπεδο της πρόληψης και της εποπτείας και ελέγχου αδειών στο επίπεδο των βιομηχανιών. Το ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η προληπτική ρύθμιση στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην αντιμετώπιση θεομηνιών και ανθρωπογενών καταστροφών. Χρειάζονται λύσεις για διασυνοριακά προβλήματα σε αυτό το επίπεδο και ένταση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα από μια θύελα αλλά επίσης και από μια χώρα που όπως άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διμερείς συμφωνίες που έγιναν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό αμοιβαία και από κοινού μεταξύ μας και ομάδες σωστικές. Η προσπάθεια προστασίας λοιπόν είναι ε, σε αυτό το σκέλος εθνική υπόθεση και η ανάγκη ανάγκες ε, ε, μιας χώρας ε, σε σχέση με μια άλλη χώρα και τις δικές της ανάγκες πρέπει να συντονίζονται και να συμφωνούνται στις δράσεις ιδιαίτερα προσεκτικά. Τα κονδύλια είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλά τα οποία απαιτούνται. Σε αυτή την περίοδο περικοπών δεν ανταποκρίνονται αυτά τα μέτρα στην κανονική τάση που θα έπρεπε να είχε ακολουθηθεί. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ευρωπαϊκή Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο έμεινε ε, πιο, κοντά από τις προσδοκίες που είχαμε. Δεν μπόρεσε να τις υλοποιήσει στο επίπεδο της πρόληψης να πάμε τόσο μακριά όσο θα ευχόμαστε. Είναι προφανές ότι η συμφωνία που επετεύχει έχει πολύ θετικές πτυχές βέβαια, διότι διευρύνει το πεδίο της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο στις θεομηνίες, που πλήττουν τους πολίτες μας αλλά επίσης και στο περιβάλλον ή τις ε, πτυχές ε, της ε, πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και επίσης ο σεβασμός των αρχών της επικουρικότητας. Μόνο με έτοιμα κράτους μέλους θα είναι δυνατόν να υπάρξει μια παρέμβαση με βάση αυτό το μηχανισμό. Δεν είναι ας το πούμε έτσι ένας μηχανισμός που αυτόματα παρεμβαίνει κατά της βούλησης των κρατών μελών. Και έτσι λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέσο έκφρασης αλληλεγγύης Είδαμε μια σημαντική αύξηση ουσιαστικά των καταστροφών που τις αποκαλούμε φυσικές καταστροφές ή θεομηνίες αλλά που πολύ περισσότερο συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές και με τον τρόπο που ληστεύει, καταλυστεύει το περιβάλλον ο καπιταλισμός και πλήττει το περιβάλλον και τους ανθρώπους από αυτή την αχόρταγη ληστρική του δίψα του καπιταλισμού. Και όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πλήττονται από αυτές τις καταστροφές είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κατεπίγουσα απάντηση, αποτελεσματική απάντηση προς όφελος των πληττόμενων πολιτών. Ε, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Ε, επιθυμούμε να μην υπάρξει καμιά πρόθεση να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς και στόχους αυτή η δράση. Όμως πολύ πιο πέρα, πιο κοντά βρίσκεται από τις ευχές που θα είχαμε για ένα τέτοιο μηχανισμό. Το e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 Τόσο ο νέος μηχανισμός στον τομέα πολιτικής προστασίας συγχωνεύει δύο νομικές πράξεις και προσφέρει και μια απλούστευση των διαδικασιών και μια επιτάχυνση, ταχύτερη δράση της προτινόμενης ε, προσφερόμενης βοήθειας. Μια και έχουμε όλο και περισσότερο, μεγαλύτερο αριθμό θεομηνιών, καταστροφών και ζημιών, είναι πολύ σημαντικό συντονισμένα να μπορεί να δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέργειες. Πρέπει άμεσα να μπορούμε να αντιδράσουμε και με μεγαλύτερη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται και μια υπηρεσία. Πρέπει όμως να πούμε ότι συμπληρωματικά μόνο μπορεί να δράσει μια τέτοια βοήθεια στο, από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο έργο είναι των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στο έργο μας. Πολύ ο συνάδελφος Όμπερμαϊερ από τους Μέγγε Γραμμένους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προστασία πολιτικών καταστροφών έχει και τις τοπικές και περιφερικές αρμοδιότητες και ιδιομορφίες. Χαιρετίζουμε σε σχέση με τον συντονισμό να βελτιώσουμε τον συντονισμό αυτό των μέσων και των δυνατοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σκόπιμο και η πρόληψη να προωθεί, να προβλέπουμε αντί να θεραπεύουμε εκ των υστέρων. Και είναι σημαντικό να ανταλλάσσουμε βιώματα και πληροφορίες για να είμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλοχαιρετίζουμε. Να μάθουμε μέσω επιτυχίας και ερεθισμάτων και όχι λόγω του ότι αυτό επιβάλλεται από κάποιους. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ο αριθμός ε, δεδομένων ε, των, ε, της δεδομένης των φαινομένων αυτών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις από πλευράς κρατών μελών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ώστε να μην υπάρχουν στενοποί. Καθώς επίσης και το στόχο, το κόστος αποτελεσματικών ε, δράσεων πρέπει να μειωθεί ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε στο μέτρο του εφικτού αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι αυτές οι θεομηνίες, οι πολλαπλασιάζονται λόγω των κλιματολογικών αλλαγών και είναι είτε ανθρωπογενείς είτε φυσικές αλλά έχουν πάντοτε τρομερές οικονομικές συνέπειες. Στη Γαλλία υπολογίζουμε πάνω από 15.000 θύματα και 30 δισεκατομμύρια χρειάστηκαν για την αποκατάσταση των σημειών. Ο μηχανισμός λοιπόν αυτός πολιτικής προστασίας πρέπει απολύτως να απλοποιη... έπρεπε να απλοποιηθεί, ήταν επίγον να υπάρχει ένας μηχανισμός που να αντιδρά γρηγορότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκείται σε αυτοσχεδιασμούς. Ενδυναμώνουμε λοιπόν έτσι τη συνεργασία, το συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών και θα έλεγα μάλιστα επιτέλους διότι από το 2006 ο κύριος Μπαρνιέ είχε κάνει μια πρώτη τέτοια πρόταση. Πράγματι χρειάζεται αυτό το κέντρο αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Είναι σημαντικό βήμα για την καλύτερη κοινή χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτουμε. Και εδώ η Ευρώπη μπορεί πράγματι να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και να παρουσιάσει υπεραξία. Γιατί 82% των Ευρωπαίων σε δημοσκόπηση θεωρούν ότι η ενωσιακή αντιμετώπιση θα ήταν πιο αποτελεσματική από την μεμονωμένη εθνική. Ο συνάδελφος Ταμπάιτη tisztelt ευχαριστώ κύριε επίτροπε. <clears throat> βλέπουμε ότι από τις ε, θλιβερές ε, εμπειρίες ε, του πρόσφατου παρελθόντος μπορέσαμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Στην Ουγγαρία ζήσαμε την τραγωδία με την κόκκινη λάσπη που έπληξε την χώρα μας, τη μεγαλύτερη βιομηχανική καταστροφή στην ιστορία μας. Στην Ρουμανία είχαμε την καταστροφή όσον αφορά το χρυσορυχείο το οποίο οδήγησε σε σοβαρότατα ζημιές και επιπτώσεις. Πρέπει εδώ λοιπόν να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις. Συμφωνούμε τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούν, να μπορούν να γνωστοποιούν στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι το διαθέσιμο δυναμικό, ώστε η κοινή δράση να μπορεί να βελτιώνεται. Είναι αναγκαίο ένα κέντρο διοίκησης και διαχείρισης αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων να δημιουργηθεί. Επίσης να δούμε τι πρέπει να γίνεται σε σχέση με βιομηχανικά τυχήματα και το ταμείο το οποίο θα μπορεί να ε, δράσει πρέπει να είναι αποτελεσματικό Ε, Πρόεδρε, Επίτροπε, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας αυτό το οποίο σημαίνει χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει όμως χρήματα. Τα χρήματα ανήκουν στα κράτη-μέλη. Και τι κάνετε, παίρνετε τα χρήματα των κρατών μελών και μετά τα συσκευάζετε εκ νέου σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παίρνετε από τη μία και τα δίνετε από την άλλη. Πρόκειται για μια στρεβλή μεθοδολογία. Είναι μια άπελπη προσπάθεια έτσι ώστε οι πολίτες της Ένωσης να αγαπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που η δημοφιλία σε εισαγωγικά της Ένωσης έχει καταρρεύσει. Δεν θα βοηθήσετε σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμύρας κτλ. Δεν αντιμετωπίζονται σωστά, υπάρχουν καταστροφές με χιλιάδες θύματα όπως τι Φιλιππίνες και θα πρέπει εμείς σαν Μεγάλη Βρετανία βοηθήσαμε πάρα πολύ και ο Βρετανικός λαός έδωσε 17 εκατομμύρια λίρες με δωρεές και το κράτος 60 εκατομμύρια λίρες με βοήθεια παρέχοντας αεροπλάνα, τροφές κτλ. Δεν θα πρέπει να σας δώσουμε λοιπόν τα χρήματα αυτά για να τα χρησιμοποιήσετε σαν προπαγάνδα νομίζω δεν είναι στην αίθουσα, δεν τον βλέπω, οπότε θα παρακαλέσω τον ε, συνάδελφο Σνέλχαρτ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πάντα υπήρχαν φυσικές καταστροφές και θεομηνείς και θα υπάρξουν και στο μέλλον. Η δική μου εκλογική περιφέρεια επλήγει ε, με τον χειρότερο τρόπο κάτω πρόσφατο παρελθόν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να δράσει αποτελεσματικά και εδώ με διαφορετικούς τρόπους να δράσουμε. Η αναθεώρηση των μέχρι σήμερα κανονισμών και διατάξεων είναι μια καλή ευκαιρία να πετύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο αυτό. Διότι ακριβώς εδώ και αυτό η εξέλιξη των τελευταίων μηνών το κατέδειξε, έχουμε κενά που πρέπει να καλύψουμε, ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Υποστηρίζουμε λοιπόν έντονα τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Κέντρου δράση και Συντονισμού, διότι εδώ υπάρχει πραγματική έλλειψη για τη συνεργασία των περιφερειών και των δράσεων μεταξύ του. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε. Το είδαμε αυτό με προηγούμενε καταστροφέ, διότι αν είχαν ληφθεί σε σχέση με τι ποτάμιες πλημμύρε όλα τα μέτρα έγκαιρα, τότε στι εκβολέ του ποταμού οι ζημιέ θα ήταν πολύ μικρότερε. Εδώ λοιπόν η ευρωπαϊκή δράση μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, και το στην ε, γεωργική πολιτική να μπορέσουν αυτά τα κονδύλια να δράσουν ε, είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση αυτών και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και όχι μόνο την αντιμετώπιση των ε, επιπτώσεων. Ένα κενό πρέπει να αναφέρω. Πόσο καιρό κράτησε ώστε να μπορέσει από μια φυσική καταστροφή, από μια θεομηνία να διατεθούν τα κονδύλια. Χρειάστηκε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν βλέπουμε πώς επιχειρήσεις πλήττονται επειδή δεν έχουν κατανεμηθεί, δεν έχουν επιμεριστεί αυτά τα κονδύλια ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει εδώ να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πολύ γοργότερα να δρούμε για να έχουμε καλύτερο συντονισμό συνολικά και να μην πλήττονται οι επιχειρήσει και να αφήνονται με στο γκρεμό λόγω του, του ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά προσκόμματα. Ευχαριστώ. Ο πρόσφατος τυφώνας που κατέστρεψε τις Φιλιππίνες δείχνει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες θεομηνίες από ό,τι πριν. Ακραία καιρικά φαινόμενα που δημιουργούν τεράστιες ζημίες. Ξέρουμε βέβαια ότι η ένταση και η συχνότητα θα αυξηθούν, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ακριβή στιγμή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για να μπορούμε να αντιδρούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ο μηχανισμός αυτός πολιτικής προστασίας θα μας βοηθήσει για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η συμφωνία με το Συμβούλιο θα βελτιώσει σημαντικά τους τέτοιους υπάρχοντες μηχανισμούς θα αποτελέσει καλύτερη, θα καταλήξει σε καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων και της πρόβλεψης και θα μας δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης, αντιμετώπισης. Δεν είναι επιφανειακή πρόοδος, αλλά πραγματική βελτίωση με βάση την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει γαλάζια κάρτα του κ. Σνάρτομα. Διδέχεστε. E, prirodne i druge katastrofe ne poznaju granice pa tako e, obrana od... Ευχαριστώ. Η πρόληψη και αντιμετώπιση των θεομηνιών πρέπει να είναι κοινή προσπάθεια, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι θεομηνίες αυξήθηκαν σε συχνότητα ενώ τα ποσά που διαθέτει που, ο, διέθετε ο μέχρι τώρα υπάρχον μηχανισμός αντιμετώπισης ήταν ανεπαρκή. Λόγω της γεωγραφίας της η Κροατία γνωρίζει συχνά πλημμύρες το χειμώνα και πυρκαγιές το καλοκαίρι όπως στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία που να μπορεί να λειτουργεί υπό οποιασδήποτε καιρικέ συνθήκες και σε συνεργασία με χώρες που είναι ακόμη και εκτός Ένωσης η κατάσβεση πυρκαγιών στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Βοσνία, Ριζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο είναι κάτι που το έχουμε ήδη πράξει εμείς. Και γι' αυτό χρειάζεται πράγματι μεγαλύτερη χρηματοδότηση της διαμεθοριακής συνεργασίας. Ο Νάτολ θέλει να σας θέσει πληρωματική, όχι. Τότε δίνω το λόγο στην συνάδελφο Σμόλκοβα. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλές και χωριστές περιπτώσεις ε, από, αυτές τις, ε, από αυτά τα πλήγματα και βλέπουμε πώς επηρεάζουν τη ζωή των άνθρωπων μας. Ε, Είμαστε υπέρ του να υπάρξει η δράση ώστε να υπάρξει η προστασία. Η ασφάλεια και η προστασία όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίση. Διότι η τύχη δεν επαρκεί να είναι κανεί τυχερό. Η σωστή προετοιμασία μπορεί να σώσει χιλιάδε ζωέ. Μια ενισχυμένη προστασία έναντι αυτών των καταστροφών είναι σημαντική υπόθεση. Σε πολλού τομεί έχουμε την ενεργοποίηση ακριβώ αυτού του μηχανισμού πολιτική προστασία την αντιμετώπιση των καταστροφών. Ζούμε όλο και περισσότερο περισσότερες χώρες που πλήττονται από τέτοιες καταστροφές. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα στη χρήση των κονδυλίων. Ελπίζουμε από αυτό το μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών και πολιτική προστασίας να δράσουμε όλο και περισσότερο στο πεδίο τη ε, πρόληψη. Πρόληψη εντό και εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Πριν περάσουμε στη διαδικασία της οφθαλμοθυρίας θα μιλήσει ο συνάδελφος Βλάσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες, κυρία Επίτροπη, κυρίες και κύριοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τροποποίηση της νέας αυτής πρότασης για τον μηχανισμό και τον χρηματοδοτικό μηχανισμό, μηχανισμό πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτικό μηχανισμό του 2007 σε μία νομική πράξη για τις διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις για αυτή την πρόταση διαπιστώσαμε ότι ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή να εγκριθεί αυτή η πρόταση διότι πέρυσι έληξε ε, το προηγούμενο χρηματοδοτικό μέσο. Στόχος ποιος είναι να απλουστευτούν διαδικασίες, να πλουστευτούν οι διεργασίες για να υπάρχει συγχρηματοδότηση όσον αφορά την προστασία και να διασφαλίζεται ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε έκτακτες περιπτώσεις έναντι ε, περιπτώσεων που συμβαίνουν σε τρίτα κράτη. Επίσης η γραφειοκρατική επιβάρυνση πρέπει να μειωθεί και αυτή, να συρρυκνωθεί. Υπό το πρίσμα της Περιφερειακής Επιτροπής θα ήθελα να αναφέρω επιπλέον ότι οι κύριες προϋποθέσεις της Προστασία εναντί τέτοιων καταστροφών πρέπει να είναι ότι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο θα πρέπει να παρέχεται η προστασία αυτή. Στι τοπικέ αρχές, περιφερειακές αρχές που πρέπει να εμπλέκονται. Διότι αυτές είναι εκείνες που έχουν την λύση έτοιμη νωρίτερα. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και πρώτα ε, θα καλέσω τον συνάδελφο Ματούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι η εμπλοκή των τοπικών αρχών είναι καθοριστική όταν θέλουμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που παρουσιάζει η πολιτική προστασία. Και γι' αυτό οι περιφέρειες θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα σε σχέση με τις συνολικές ε, συλλογικές παρεμβάσεις η ομοιογένεια των τρόπων με τους οποίους παρεμβαίνουν οι διαφορετικές υπηρεσίες καθορίζει την ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες. Η αυξημένη κινητικότητα είναι απαραίτητη μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών οδών. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την απόκριση στις ανάγκες Η επιτόπου λοιπόν παρέμβαση με τη βοήθεια εθέλοντων, ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, είναι κάτι το οποίο και αυτό με τη σειρά του βοηθά. Ο εθελοντισμός ε, και οι εθελοντές σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες βοηθούν πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, στην... πρέπει να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην ξεχνάμε την αποτελεσματική δράση. Η πρόληψη έχει κύριο ρόλο στην αντιμετώπιση καταστροφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνωρίζει στην πρότασή της αυτό. Αναφέρεται και μέχρι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σεπτεμβρίου 2010 που ήμουν εγώ συντάκτης του για μια κοινοτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση θεομηνιών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ε, πρέπει εδώ να προαρθούν όλες οι συστάσεις που περιέχονται σε εκείνο το ψήφισμα. Δημιουργία ενός σωστού πλαισίου για την χρηματοδότηση της πρόληψης των καταστροφών αντιμετώπιση των καταστάσεων κινδύνου όσον αφορά για παράδειγμα την, τις ακτές, τα δάση, τις ε, υδρογραφικές λεκάνες, ε, τις ζώνες που έχουν ε, κανονικότερο, πυκνότερο πληθυσμό εναντί άλλων. Όλα πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τομέα και η πρόληψη. Αναμένουμε επίσης μια αναθεώρηση του κανονισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης που θα επιτρέπει κινητοποίηση πιο ελαστική και πιο αποτελεσματική έγκαιρα. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος Γεωργίεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση για τα σχόλια τους. Τέσσερα θέματα να διευκρινίσω. Πρώτον, για αυτήν την ε, νομοθετική περίοδο προσπαθούμε να συλλάβουμε την επιθυμία των πολιτών μας. 9 στους 10 Ευρωπαίους μας είπαν ότι θέλουν να συνεργαστούμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε απειλές που απειλούν τα δικαιώματά τους στην ιδιοκτησία τους, την ίδια τους τη ζωή. Δεύτερον, Ε, αυξάνουμε αν θέλετε το επίπεδο αλληλεγγύης εκεί όπου χρειάζεται, εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ε, το 90% των φυσικών καταστροφών είναι τοπικής μορφής, οπότε εκεί η αλληλεγγύη δεν παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά για το 10% που ξεπερνούν τις χώρες μας ε, ή και τρίτες χώρες, τότε αυτή η επίδειξη αλληλεγγύης κάνει τη διαφορά λιγότερα θύματα, μικρότερες ζημίες. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να ελέγξουμε ε, και τις ίδιες τις ικανότητες ε, των δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Όταν συνεργάζονται, όταν εκπαιδεύονται μαζί και όταν αναπτύσσονται μαζί είναι πιο αποτελεσματικές οι δυνάμεις αυτές. Να πω επίσης ότι εμείς ελέγχουμε και το θέμα της αλληλεγγύης μέσω των ποσών που συγκεντρώνονται για λόγους αλληλεγγύης έτσι ώστε αυτά τα μέσα να χρησιμοποιηθούν σωστά μέσω των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Τρίτον, ε, εδώ σεβόμεθα την αρχή της επικουρικότητας. Είναι εκ των κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίθετο. Και είμαι ευγνώμων σε όλους αυτούς οι οποίοι αναγνώρισαν αυτήν την ιδιότητα ότι δηλαδή κάναμε μια καλή δουλειά σε συνεργασία με, το κράτος μέλος, με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλος, ε, είναι η αποτελεσματικότητα του κόστους, αν θέλετε, αυτών των παρεμβάσεων. Ε, χρειάζεται μια κουλτούρα ε, γνώσης των συστημάτων αυτών. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μέλλον λόγω των κλιματικών αλλαγών με πολλές φυσικές καταστροφές και γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε καλύτερα την ασφάλεια των πολιτών. Συντονισμένη ανταπόκριση, ε, πράγματι το σύνολο όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι μεγαλύτερο από την απλή μορφή συνδυασμού των επιμέρους ικανοτήτων. Ελπίζουμε λοιπόν να εφαρμοστεί το ταχύτερο η προτινόμενη νομοθεσία και ε, το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής θα είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ την κυρία Γεωργίευα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Γκαρντίνη. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και την Επίτροπο. Έχουμε να κάνουμε με κάτι σημαντικό. Μιλάμε για αλληλεγγύη, για ευρωπαϊκό πνεύμα, για πολίτες οι οποίοι ακόμα και σήμερα ζητούν ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη Ευρώπη κάτι το οποίο σπανίζει τον τελευταίο καιρό. Και μιλάμε και για μια πολιτική προστασία που δουλεύει. Στη χώρα μου αυτές τις μέρες, στη Βενετία, ξεκίνησε χθε και θα κρατήσει τέσσερις μέρες η εξέλιξη μιας πανευρωπαϊκής άσκησης στην οποία συμμετέχουν ομάδες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Εστονία, την Ουγγαρία και την Ιταλία φυσικά. Μιλάμε για έναν ισχύοντα μηχανισμό ευρωπαϊκό, λειτουργικό Επί τη βάση της εμπειρίας που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα θέλουμε να τον καταστήσουμε πιο αποδοτικό. Τα χρήματα που θέτουν στη διάθεσή μας τα κρατημέλη είναι λίγα, ιδιαίτερα για τον τομέα της πρόληψης. Θα έπρεπε ιδιαίτερα στην πρόληψη να επενδύσουμε δισεκατομμύρια, γιατί η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την εκ των υστέρων παρέμβαση μετά την καταστροφή. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η 16η επέτειος ε, της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού στο Φριούλ και την περιοχή της Βενετίας. Αναγνωρίζεται η προσπάθεια που έχουν κάνει οι τοπικοί πληθυσμοί και ο Επίτροπος Τζαμπερλέτη. Ε, πράγματι αν βλέπατε ε, τι συζητούσαμε θα καταλαβαίνατε γιατί συζητάμε. Μιλάμε για μια κοινότητα που μετά από 40 χρόνια από μια ε, ισχυρή σεισμική δόνηση εξακολουθεί να φοβάται, δημιουργούνται πάντα προβλήματα σε μια περιοχή ενός εκατομμυρίου 200.000 πολιτών. Οι εθελοντές και το ποσιστοκοποιήσαμε τον τελευταίο καιρό έχει προσφέρει πολλά, έχουν προσφέρει πολλά που έχουν προσφέρει το ισόποσο πάνω το από 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει ότι αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα, ότι ε, πιστεύουν στην αλληλεγγύη, ότι παρόλους τους φόβους και τα προβλήματα μπορούν να βοηθήσουν το έδαφος τους, στην περιοχή τους, να την καταστήσουν πιο ανθεκτική, πιο ισχυρή, πιο θωρακισμένη και έτσι να τη μεταφέρουν στα παιδιά τους και στους επιγόνους τους. Έτσι λοιπόν εδώ θα βοηθήσει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η ψηφοφορία που θα γίνει σήμερα φαίνεται κάτι το ασήμαντο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία την οποία έχουμε μαζί διανύσει και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κρυσταλίνα Γεωργίευα για το πάθος και την καρδιά. Η ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Γκαρντίνη θα γίνει σήμερα στις 11.30 και η συνεδρίασή μας διακόπτεται έως τότε. Θα επανέλθουμε στις 11.30 για την ψηφοφορία.